Απουσιάζει η κυρία Τόγια. Άρα η κυρία Καρδίνη, η επόμενη. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να σας πω και σας παρακαλώ να προσέξετε διότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που συνέβη και αναφέρθηκε στον Ιταλικό τύπο τις περασμένες ημέρες μάθαμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής στο δεύτερο Wikileaks, Data Datagate, ε, από τον τότε πρόεδρο του Σίλβιο Μπελουσκόνη το 2011 και πριν τον παρακολουθούσε αυτόν και τους συνεργάτες τους. Οπότε μετά τη Γερμανία, μετά τη Γαλλία είδαμε και η Ιταλία παρακολουθεί το από σύμμαχο. τα λόγια που είπε ο πρόεδρος Σούλτς που χρησιμοποίησε τις προάλλες σε ένα Ιταλικό πρόγραμμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό διότι δεν είναι δίκαιο στις συμμαχικές χώρες να παρακολουθούνται η κυβέρνηση τη Ιταλία το επαληθεύει και το συζητάμε με τι ΗΠΑ. Θα θέλαμε θα πρέπει να γίνει ένα και στο Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τι δραστηριότητε, τη κατασκοπή που γίνεται ει βάρο τη ε, Ευρώπη. Είχε λήξει η έρευνα το Μάρτιο του 2014. Δεν θέλουμε να είμαστε ύποπτοι και να υπάρχουν σκιέ μεταξύ συμμαχικών χωρών. Και ζητάμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να μα βοηθήσει ούτω ώστε να ρίξουμε φω. Ε, διαφορετικά ε, γνωρίζετε ότι και ευαίσθητες εμπορικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν ε, υπάρχουν σημαντικές πτυχές που αφορούν αυτή τη συλλογή πληροφοριών. Ευχαριστούμε, ακούσατε αυτά που είχατε να πείτε. Η κυρία Τόγια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω και από τη δική μα πλευρά ότι οι ειδήσει που μάθαμε από τον τύπο και αποκαλύπτουν κατασκοπιστικές δραστηριότητε από πλευρά διαφόρων οργανώσεων ε, των ΗΠΑ κατά ε, των ευρωπαϊκών χωρών είναι πάρα πολύ ενσυχητικέ ειδήσει και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε καθησυχώντα, διότι, ε, διότι παντού γίνεται αυτό. Υπάρχουν χώρε και σχέσει μεταξύ χωρών που πρέπει να διέπονται από σεβασμό και διαφάνεια όσον αφορά τι αμοιβέ αυτονομίε και θα πρέπει να πολεμήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ακούσαμε αυτά που μας είπατε και θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα είναι η έκθεση του κύριου Σπάσκη. Το λόγο ζήτησε ο εισηγητής μας, ο κύριος Σπάσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Σύμβαση της Χάγης του 1965 δημιούργησε ένα σύστημα που απλουστεύει την ανταλλαγή ε, εγγράφων και δικογράφων μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, ε, διευκολύνει τα δικαστήρια και τη δικαστική συνεργασία σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου. Η σύμβαση της Χάγης ε, έχει αποδειχθεί χρήσιμη. Μάλιστα την ε, εφαρμόζουν 25 χώρες μέλη και η Αυστρία και η Μάλτα επίσης εκδήλωσαν την επιθυμία να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή. Έγινε εκτενέστατη συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό και τα δύο κρατημέλη, Αυστρία και Μάλτα, έλαβαν την εξουσιοδότηση να προσχωρήσουν στην σύμβαση. Θα ήθελα να παρακαλέσουν, του αδέλφου να υπερψηφίσουν τη σύσταση, ώστε να μπορέσουν και η Αυστρία και η Μάλτα να προσχωρήσουν στη σύμβαση τη Χάγη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Με ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα, η έκθεση της κυρίας Βανιούενχόιζεν με ονομαστική κλίση, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τρίτη έκθεση του κυρίου Σδεχόφσκι, με ονομαστική κλίση και αυτή, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Επόμενη έκθεση του κυρίου Μπέκερ. Εδώ θα κρατήσει πιο πολύ ψηφοφορία. Πρώτα τροπολογία 177. Διανατάσσεω τη χειρός. Παρακαλώ, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Η 177 τροπολογία. 181 και 183 τώρα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτονται. Τροπολογία 178. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 179. Ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 177 διανατάσεις της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 180 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. Τροπολογία 177, διανατάσεις της χειρός, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182, διανατάσεις της χειρός, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Διανατάσσεω στις χειρώσεις τη πρόταση τη Επιτροπή. Ποιο είναι υπέρ, κατά. αποχές Εγκρίνεται. Και το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σδεχόφσκι. Έκθεση της Αρνές τώρα, τροπολογία 16, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία από την αρμόδια ουσία επιτροπή, ε, συνολική. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 13, διανατάσσεως τη χειρό, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αν θέλετε, για την τροπολογία 13, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 5 και 12 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 6. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 7 και 14. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψυχοφορία. Τέλος. Απορρίπτονται. Τροπολογία 8. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 δυνατά στους χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 με τα χέρια πάλι Α, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 10. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 11 και 15. Διανατάσεις χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 11 και 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται, συγγνώμη. Πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ο κύριος Λάγκε ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής και εγώ λυπούμεθα ότι το κείμενο ε, το οποίο είχαμε διαβαγματευτεί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν εγκρίθηκε χωρίς τροποποίηση. Ήταν ε, άμεσα μέτρα για να υποστηρίξουμε την, την Για να μην χάσουμε ακόμη περισσότερο χρόνο θα ήθελα να ζητήσω να αναβληθεί η τελική ψηφοφορία για να ξεκινήσουμε αμέσως τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο για να βρούμε σύντομα μια λύση και να δώσουμε σύντομα βοήθεια στην Τινησία. Okay. Μάλιστα. Η, η συγγήτρια ζήτησε να αναβληθεί τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ να ψηφίσουμε επί του αιτήματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται το αίτημα της αναβολής. So we go to... Uh, by... Περνάμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Ζδεχόφσκι. Ψηφίζουμε το ψήφισμα ολόκληρο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Ροντρίγκες. Τροπολογία 6. Ένα διαδικαστικό. Ε, γρήγορα. Μου είπαν οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου ότι έγινε ένα λάθος όσον αφορά την τροπολογία 13. Εμείς είχαμε βάλει σαφώς την αναφορά στην Τραπεζική Ένωση και αλλά στη μεταρρύθμιση εθνωτική της Απεζικής Ενώσεως. Αντί μπήκε το Banking Union. Θέλουμε λοιπόν την τροπολογία χωρίς τις λέξεις Banking Union, την Τραπεζική Ένωση. Η νομική υπηρεσία θα κάνει τις ε, αναγκαίες διορθώσεις, λέει Πρόεδρος. Τροπολογία 6, ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο δυνατά ισχυρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25, δυνατά ισχυρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας απορρίπτεται 26 ανατάσσω στη σειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 27 Διανατάσταση της χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 7 Διανατάσταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 δυναμωστικής πληροφορίας που άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ναι, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9 του αρχικού κειμένου. Διανετάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 διανομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα, δυνατά χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δυνατά χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές μάλλον. Κατά. Λέει Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, δεν θα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Δεν θα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Διανομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. απορρίπτεται. Παράγραφος 12 του αρχικού κειμένου διανατάσσει χειρός υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 29 διανατάσσει χειρός υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Παράγραφος 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διανατάσσει χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα διαντάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 διανομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται πέρας απορρίπτεται Τροπολογία 16, Διανομαστική ψηφοφορία. που άρχεται. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31, διανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 19 διανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 διανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 33 διανομαστικής ψηφοφορίας παρέρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Διαντάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. διανομαστική ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. απορρίπτεται. Παράγραφος 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, διαντάσεις χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, διανομαστικής ψηφοφορίας, άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, διανομαστικής ψηφοφορίας, πάρχεται, Πέρας. τροπολογία 18. Δυνατάς ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Διονομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24. Δυνατάς ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 35. Δυνατάς ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Διανομαστικής ψηφοφορίας πάρχεται. Πέρας αυτής. απορρίπτεται 26 παράγραφος 26 δυνατά συγχυρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 διανομαστικής ψηφορίας που άρχεται πέρας απορρίπτεται τροπολογία 2 Ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Διονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Δυνατάς ισχυρός υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται παράγραφος 27 δύο τμήματα πρώτο τμήμα δεν τα χειρός υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα δεν τα χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 36, Διανατάσταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28, σε τρία τμήματα, διανομαστικής ψηφοφορίας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, διανομαστικής ψηφοφορίας, που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, διανομαστικής ψηφοφορίας, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21, διανομαστικής ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 30. Δυνατά στο σχηρός πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Διανομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 32. Διανατάς χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Διανομαστικής πληροφορίας. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38 διανομαστικής ψηφορίας που ξεκινάει τέλος απορρίπτεται τροπολογία 38 37 συγγνώμη λέει πρόεδρος 39 διονομαστική ψηφορία της χειρός υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Παράγραφος 35 δυνατά στις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά παράγραφος 36 δυνατά στις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 38. Ε, διανατάσσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 40. Διανατάσσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 43. Διανατάσεως υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 46. Διανατάσεως υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 47. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Διανατάσσεω υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 48. Διανατάσσεω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 51 διανατάσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 διανατάσεως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 24 διανατάσεως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη I διανατάσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και να ψηφίσουμε συνολικά το ψήφισμα διαναστικής ψηφοφορίας άρχεται πέρας εγκρίνεται και συγχαίρω τον συγητή. Έκθεση της κυρίας Ριμπέιχου. Τροπολογία 1. Διανατάσσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραγράφος 6. Δύο τμήματα. Διανατάσεως. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Διανατάσεως. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Διανατάσσεως υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Διονομαστικής άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 20 λοιπόν. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται, πέρας, Απορρίπτεται. Παράγραφος 25. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, καλά έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Διανατάσιος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 39. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 41. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Έλεγχος. Άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Παράγραφος, α, συγγνώμη, δεύτερο τμήμα, ε, διανατάσσεως, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 42. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Διανατάσεις υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 43. Δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 53. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 59. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 62. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 64. Τέσσερα τμήματα. Ονομαστική όλα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 69. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 70. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, έλεγχος. Για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Άι. Δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ωραία, να ψηφίσουμε το ψήφισμα συνολικά, ονομαστική ψηφοφορία. vote is open. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια. Ωραία, περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Τέιλερ Παράγραφος 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 35. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται οι, τροπολο... παράγραφοι 46 και 52 καταπίπτουν και μάλλον ε, ε, οι 52 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Πάμε στην τροπολογία 12 για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Τινησία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 11 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 13 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 4. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία... Α, καλά. Αφού επιμένετε ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 7, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο 44. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 57. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 58 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα της, τροπο... της παραγράφου 59. Διανατάσεις χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται και το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται περνάμε στην έκθεση της κυρίας Καμπεσόν, Καμπεσόν Ρουής τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά άποχες Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το πρώτο τμήμα δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό τροπολογία 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και 11 ποιος είναι υπέρ. Ας κάνουμε όμως πρώτα έναν ηλεκτρονικό έλεγχο για την παράγραφο 29, την τροπολογία 10 δηλαδή, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 10. Τέλος απορρίπτεται. Και τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ολόκληρο το ψήφισμα τώρα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια την εισηγήτρια. Έκθεση του κυρίου Μαριά τώρα, τροπολογία 6, διανατάσσεως της χειρός, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 6, σε δύο τμήματα, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 6. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος απορρίπτεται. Παράγραφος 15, πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Ηλεκτρονικό έλεγχο για το τρίτο τμήμα τη παραγράφου 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα τη παραγράφου 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία το σύνολο του ψηφίσματος, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μαριά και έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα μιλήσω ελληνικά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ το Σώμα για την υπερψήφιση της έκθεσης η οποία περιέχει αρκετά σημεία κριτική στη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τρόικας. Φυσικά υπάρχουν πτυχές στην έκθεση, όπως σε κάθε έκθεση, που δεν εκφράζουν τον εισηγητή, όπως το τρίτο μέρος της παραγράφου 15. Για όλα αυτά θα καταθέσω γραπτά τις απόψεις μου στα πρακτικά. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έναρξη διαπραγματεύσεως ε, ε, ε, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τροπολογία 8 δυναμαστικής ψηφοφορίας. Άρχεται ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Πάμε στην τροπολογία 10. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Εντάσσεως χειρός. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφορία, Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G. στις χειρός υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5. Η ανατάσσος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Το ψήφινο συνολό τη ονομαστική πληροφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε την καταγραφή καταχώρηση ζώων συντροφιά στα κάτι μέλη. Είναι κοινό ψήφισμα που στηρίζεται από έξι ομάδες, τοπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τοπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τοπολογία 1 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εταιρική σκέψη G. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεν ήταν ξεκάθαρη εικόνα. Θα ψηφίσουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη. Ήτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σαφέστατο αυτό Πάμε στην τελευταία ψηφοφορία για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Ο κύριος Πρέντα θα ήθελε να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να εκφράσω για την ψηφοφορία στις 4 Φεβρουαρίου, την απογοήτευσή μου, και διακόπτω το μικρόφωνο το μιλητή. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Κύριε Πρέντα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι η ομάδα μας είναι κατά της τροπολογίας που κατετέθη από τους σοσιαλιστές, φιλελευθέρους και άλλους που καθιστά το ψήφισμα πολύ ε, ανισόρροπο θα έλεγα. Είναι ένα κείμενο που υποστηρίζει τη Σαουδική Αραβία με υπερβολικό τρόπο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε σε όλους τους φορείς της περιοχής συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Πήγε με αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία που συναντήθηκε με τον Βασιλιά και πολιτικές ομάδες που πρότειναν την τροπολογία δεν υποστήριξαν τη θέση αυτή όταν ήταν εκεί. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα πράγματα στη Σαουδική Αραβία και άλλα εδώ. Κύριε Πρέντα, λέει πρόεδρο, δεν θα πρέπει να διεξαχθεί η συζήτηση τώρα, αλλά η ψηφοφορία. Συζητήθηκε αυτό ήδη στο Στρασβούργο. Διαδικαστικό. Ο κύριος Κάρμπερ. Κύριε Πρέντα, ήθελα να πω το, ότι καθυστερήστε και η ψηφοφορία στις 4 Φεβρουαρίου, το θέμα αυτό η ψηφοφορία για να, ε, για να είμαστε ευγενικοί διπλωματικά κλπ. Έκτοτε πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα εκφράζουν την αηδία τους. Πέθαναν περισσότεροι, έχει διαδοθεί η χολέρα, ε, οι υποδομές έχουν επιδεινωθεί και αυτό είναι κρίμα που καθυστερήσαμε τόσο. Από τις 4 Φεβρουαρίου πρέπει να ψηφίσουμε, λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε, λοιπόν, πρόταση ψηφίσματος της ομάδας του ECR πρώτα. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το κοινό ψήφισμα που στηρίζεται από έξι ομάδες, πρώτη είναι η τροπολογία παριθμών 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήταν σαφέστατη η εικόνα. Παράγραφος 6 Καλώς, εντάξει, θα ελέγξουμε. Τροπολογία 3 θα γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6 του αρχικού κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 1, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ψηφίσατε, πρέπει να ελέγξουμε υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Έλεγχος, όχι ονομαστική ψηφοφορία. Γιατί είδα ελάχιστα χέρια να σηκώνονται. Πέρα. Εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική σκέψη. Νη. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Ενεκριθεί. Now we come to the explanation. Πάμε στις επεξηγήσεις ε, ψήφου. Εκείνοι που θέλουν να πούν κάτι θα παρίστανται για να πάρουν το λόγο. Ήρθε η ώρα για την επεξήγηση ψήφων. Καταρχάς, έχουμε την έκθεση Μπέκερ, η πρώτη επεξήγηση ψήφου, η κυρία Μορβάη. Κυρία Μορβάη, έχετε το λόγο. Λυπάμαι πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπαινοβγαίνει κόσμος στην αίθουσα. Υπάρχουν πολλές κουβέντες σαν ένα καφενείο. Αυτό είναι προσβολή κατά των ψηφοφόρων, κατά των